President, wieder aufgenommen. Γεια σα. Καλησπέρα σα Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Έχετε τα πρακτικά τη χθεσινής συνεδρίασης στη διάθεσή σα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει, Αν όχι, εγκρίνονται τα χθεσινά πρακτικά. Ο πρόεδρος ε,